pani przewodniczącej! witam państwa bardzo serdecznie. wznawiam. επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μα. τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης και τα εγκριθεί είναι ήδη διαθέσιμα. Πρώτο θέμα της ε, η ημερησία διάταξη είναι συζήτηση για περιπτώσει παραβιάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Πρώτο